Και η επόμενη συνεδρία θα λάβει χώρα αύριο, 4 Φεβρουαρίου 2014. Η ημερήσια διάταξη έχει δημοσιευτεί και μπορείτε να τη βρείτε στο, στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εδώ ολοκληρώνω τη σημερινή μας συνεδρίαση.